Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση τη κυρίας Άννα Γκόμες για το θέμα της Σαουδική Αραβίας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητρία για 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Σαουδική Αραβία στην ε, Μέση Ανατολή και σε παγκόσμιο επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο οικονομικά σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, παρά το γεγονό ότι η Σαουδική Αραβία επίσημα ε, δεν ε, είναι πάντα υπέρ της καταπολέμησης ε, της τρομοκρατίας, γιατί ο χαμπισμός και οι ακραίες, τα ακραία κινήματα χρηματοδοτούν την τέτοιες δράσεις σε πολλές περιφέρειες, σε πολλές χώρες. Μπορεί να υπάρχει διαφορετική βούληση στο ΡΙΑΤ, αλλά οι συνέπειες ήταν τραγικές στη Συρία, στην Αίγυπτο, στο Μπαχρέιν, στη Λιβύη, στο Μαλί, στο Ιράκ, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν. Προκάλεσε τριβές εθνοτικές. Δεν μπορούμε λοιπόν να σιωπήσουμε σε ό,τι αφορά τα προβλήματα αυτά σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις μας με τη Σουδική Αραβία. Προβάλλεται συχνά η οικονομική διάσταση και Βραχυπρόθεσμα θέματα ασφαλείας. Φυσικά είναι μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου, σημαντικός παράγοντας στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μέλος του G20, αγοραστής όπλων. Αλλά υπάρχει και στρατηγική διάσταση στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σοδικής Αραβίας. Υπάρχουν θέματα σύγκλησης αλλά και προβλήματα. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να φλούμε. Και αυτό ασφαλώς έχει να κάνει και με την καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Θέλουμε να συνεπάρχουν κουλτούρες και πολιτισμοί με ειρηνικό τρόπο. Πρόκειται για μια αυταρχική μοναρχία. Αλλά όλα αυτά έχει και διεθνείς υποχρεώσεις στη Σαουδική Αραβία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των γυναικών. Το περασμένο Νοέμβριο παρευρέθηκα στην Σαουδική Αραβία και είδα με τα ίδια μου τα μάτια ότι υπάρχει μια καταφανής ε, παραβίαση και διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία. Πρόσφατα ε, εκλέχθηκαν το 30 γυναίκες στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Σούρα και προσεχώς μόνο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές. Υπάρχει το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών. Πάντα είναι κάποιος άνδρας αυτός ο οποίος εκπροσωπεί από την οικογένεια τις γυναίκες. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας. Διακριτική μεταχείριση λοιπόν παντού κατά των γυναικών. Στην οικονομία, πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, στη δικαιοσύνη. και δεν μπορούν οι γυναίκες να οδηγούν στη Σαουδική Αραβία. Η μοναδική χώρα στον κόσμο που συμβαίνει αυτό δεν είναι όμως μόνο οι γυναίκες που υπόκεινται διακριτική μεταχείριση. Πολλά ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται σε ό,τι αφορά τους ε, θρησκευτικού δίκαστες, δεν υπάρχει ποινικό κώδικας γραπτός και στα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις θανατικές καταδίκες, βλέπουμε ότι καταδικάζονται ακόμα και ανήλικοι. Γίνονται συλλήψεις, βασανιστήρια ανθρώπων, σωματικά βασανιστήρια και σωματικός σοφρονισμός καταπατώνται τα δικαιώματα των μεταναστών θα ήθελα να αναφέρω και το σύστημα και την πρακτική. Χαρακτηριστικά για τη χώρα και είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Είναι πολύ νεαρός ο πληθυσμός τη Σαουδικής Αραβία και συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Καταπνίγεται λοιπόν από τα αναχρονιστικά αυτά συστήματα. είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Να ελεγχθεί το πρινικό πρόβλημα του Ιράν και το Ριάτ μπορεί να παίζει, να παίξει εδώ πέρα σημαντικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Και ίσως έτσι θα πάυσουν και αυτοί οι πόλεμοι στη Συρία και ίσως θα σταθεροποιηθεί και το Πακιστάν και το Ιράν. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στη συζήτηση. Ολοκληρώνει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Παίρνουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης την έκθεση του κυρίου Κόουαλ σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό